ευχαριστώ τις διάφορες χώρες που ζήτησαν και προσφέρθηκαν να μας βοηθήσουν σε μια δύσκολη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα πρακτικά της 29ης Οκτωβρίου είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν κάποια σχόλια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ο Πρόεδρος των βουλευτών, ως μάλλον, ως, ως επικεφαλής των βουλευτών τη S5, επιθυμώ να πω εξ ονόματό μα και νομίζω ότι μπορώ να το πω και εξ ονόματο ολόκληρου του Κοινοβουλίου ότι η θλίψη μα είναι βαθιά για τον Helmut Schmidt, πρώην καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, μεγάλο πολιτικό, μεγάλο δημοκράτη, μεγάλο Ευρωπαίο. Παρακαλώ το Προεδρείο στο Στρασβούργο στην επόμενη περίοδο συνόδου να τιμηθεί η μνήμη του και το ζητώ από τώρα έτσι ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί η εκδήλωση αυτή με τον κατάλληλο τρόπο. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. And thank you for your words. Um, σας ευχαριστώ για τα λόγια σας αυτά. Σε σχέση με την έγκριση των πρακτικών της 29ης Δεκάτου, επειδή δεν υπάρχουν σχόλια μπορώ να θεωρήσω ότι εγκρίνονται. Κύριε Βερχόφστατ. Κυρία Πρόεδρε, διαδικαστικό, αν μου επιτρέπετε. Χθες ακούσαμε τον Βρετανό Πρωθυπουργό να εκφωνεί ομιλία στο Chatham House και έστειλε επίση επιστολή στον Ντόναλτ Τούσκ. Είναι προφανές ότι οι αλλαγές που ζητεί ο κύριος Κάμερον είναι σημαντικές. Υπάρχουν ταυτόχρονα και άλλα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καλούμε να αναλύσουμε. Ως γνωρίζετε, ζητήσαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι παρόν ο ε, Πρωθυπουργό κ. Κάμερον να έλθει ενώπιον μας και να εξηγήσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα αιτήματά του. Πρόκειται για τον βωμό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Η δική μου επιθυμία το αίτημα που εκφράζω είναι να προσκληθεί ο κύριος Κάμερον για να προσέλθει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πράγματι θα ζητήσουμε πληροφορίες από τον πρόεδρό μας ε, για το ερώτημά σας. Έχει σταλεί πράγματι μία πρόσκληση και θα περιμένουμε να ενημερωθούμε. Άλλο διαδικαστικό, ο κύριος Δεγκράφ voorzitter eh, eh, σήμερα είναι η επέτειος της 11ης Νοεμβρίου, του τέλους δηλαδή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Ε, γνωστά τα τραγικά γεγονότα της περίοδου εκείνης που έπληξαν πολλές χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακόπτει η Πρόεδρος, φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την διερμηνία των λόγων σας. Προς κάποια γλώσσα δεν ε, ακούγεται η μετάφραση. Μπορώ να συνεχίσω στα αγγλικά, λέει ο κ. Δεγκράφ. Θέλετε να συνεχίσω στα αγγλικά? Μια στιγμή, περιμένετε παρακαλώ κύριε. Μπορείτε να συνεχίσετε. Ε, έλεγα λοιπόν κυρία Πρόεδρε ότι σήμερα είναι η Νοεμβρίου, δηλαδή η επέτειος του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου πολέμου που σημείωσε με τραγικό τρόπο την ιστορία της Ευρωπαϊκής Επίρου και με εκατομμύρια νεκρούς. Υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις οποίες η σημερινή ημέρα είναι και η μέρα εθνικής επαιτίου όπου δηλαδή αναλογίζεται κανείς τη μνήμη των νεκρών. Και όμως σήμερα διεξάγουμε εδώ συνεδρίαση και ένας αριθμός ε, των Ευρωβουλευτών δεν μπορούν να είναι παρόντες ή παρούσες διότι ε, ε, βρίσκονται στις χώρες τους για την επέτειο. Λυπούμε λοιπόν που γίνεται σήμερα η συνεδρίαση αυτή ενώ θα μπορούσε να γίνει σε άλλη ημέρα. Δεύτερον, ως πρόεδρος μπορείτε να συμβάλλετε στην ανάμνηση της μνήμης των νεκρών. Thank you for bringing this attention. I think... Σας ευχαριστώ που το φέρατε στην ε, προσοχή μας. Ακούγοντας αυτά τα οποία είπατε δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει. Και θα στείλουμε το μήνυμά σας στον Πρόεδρο και στο γραφείο του Πρόεδρου. Να πω επίσης ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής ε, για το βραβείο Λουξ. Υπάρχουν τρεις ταινίες, το Mediterranean, το Mustang και το Γιούροκ, τα οποία μπορείτε να βρείτε ε, στις προβολές οι οποίες θα γίνουν ή ακόμα και ε, ζητώντας ένα DVD. Είναι μια ειδική μέρα σήμερα γιατί για πρώτη φορά ένα από τα κινηματογραφικά αυτά έργα, το «Μεντιτεράνια», θα προβληθεί ταυτόχρονα σε οκτώ πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Γιώνας Καρπινιάνο, θα είναι μαζί μας εδώ στις Βρυξέλλες. Α, κυρία Κώστα, δεν σας είδα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που υπενθυμίσατε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό συμβάν, τη σημασία που έχει δηλαδή για τους ε, ε, παλαιούς και νέους ευρωβουλευτές που δεν γνώριζαν ίσως ε, τη διαδικασία αυτή να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία για αυτά τα έργα, τα κινηματογραφικά έργα τέχνης θα έλεγα κινηματογραφικά έργα που έχουν ήδη προβληθεί σε κινηματογραφικά φεστιβάλ αυτές τις μέρες όπως το Κάρλο Βιβάρι στην Βενετία και αλλού. Πρόκειται για τρεις ταινίες που είναι πρώτα έργα αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολύ όριμα έργα τα οποία ε, προσέχουν την έννοια της Ευρώπης και συγκεντρώνουν την προσοχή τους εκεί. Το βραβείο αυτό θα δοθεί από τον πρόεδρό μας τον κύριο Σούλτσου στον νικητή που θα επιλεγεί από μας. Πρέπει λοιπόν να ενδιαφερθούμε για το θέμα αυτό και ακριβώς το πρώτο βραβείο στην ουσία συνίσταται στο να υπάρξει υποτιτλισμός και των τριών αυτών έργων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σας ευχαριστώ κυρία Κώστα για τις επιπλέον πληροφορίες. Περνάμε τώρα στην ανακοίνωση της παρέτησης του Παύλο Ιγλέσιας και του Φερνάντο Μάουρα Μπαραντιαράν. Σύμφωνα με τον κανόνα, με τον άρθρο του κανονισμού, ε, η θέση